και ζητώ από τους συναδέλφους να ενισχύσουν ε, τις κυβερνήσεις της Πολωνίας για την, απελε... την κυβέρνηση της Πολωνίας για την απελευθέρωση του κατουμένου. Thank you. Uh, I put amendment one uh, by the committee to the vote. Those in favor. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η πρόταση όπως τροποποιήθηκε ψηφίζεται ολοκλήρου υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ο κύριος Φάβα νομίζω έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Με την άδειά σας θέλω να ζητήσω από το Συμβούλιο και μαζί με την υποστήριξη των υπόλοιπων ομάδων την